commencer sérieusement là. On a beaucoup de votes aujourd'hui. Θα ξεκινήσουμε τώρα, συνάδελφοι, γιατί έχουμε πολλές συμφορίε. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, υιοθετείτε μέσα στη διάταξη. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση της συνεδρίασης στο ίντερνετ μέσω της εφαρμογής e-meeting. που επιτρέπει και στους ευρωβουλευτές και στους βοηθούς τους ε, να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της συνεδρίασης. Έχουμε πλήρες βοήθεια καθεστώς. Να σας υπενθυμίσω τη διαδικασία. Θα ξεκινήσουμε από την ψηφορία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διασύνδεσης. Έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου, της κυρίας Βιρκούνεν και του κυρίου Τέλτσκα. Υπενθυμίζω ότι οι δύο επιτροπές, Ήτρε και Τραν, έχουν συμφωνήσει ε, να συμπροεδρεύουν οι πρόεδροι των δύο επιτροπών. Είναι πραγματικά εξαιρετική η συνεργασία με τον συνάδελφο Μπούζεκ και με τους συζητητές. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για αυτή την έκθεση θα γίνει σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα από την ε, συμβαστική CA1 έως τη συμβαστική CA17. Συμπεριλαμβάνεται δηλαδή και το άρθρο 17 εδώ. Και θα προεδρεύσω εγώ αυτή τη ψηφοφορία. Το δεύτερο τμήμα. Αρχής γενομένης από την συμβαστική τροπολογία 18 έως και το τέλος. Εκεί θα προεδρεύσει ο κύριος Μπούζεκ. Θα υπάρξει ψηφοφορία για την εντολή έναρξης των διαπραγματεύσεων. Θα περάσει απευθεία στην Ολομέλεια. Και εκεί θα αποφασίσουμε την παραπομπή στις αρμόδιες επιτροπές για την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, Ήτρε θα μπορέσει να ενημερώσει ότι η ψηφοφορία θα γίνει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στην Ολομέλεια. Να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Μπούζεκ να πει δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Μπούζεκ. Καλημέρα σε όλους. Τι ωραία καλημέρα. Ωραία. Ας ελέγξουμε ότι όλα είναι εντάξει, ότι όλοι είναι εδώ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ah, les Verts, ils ont voté en plus. Non, mais c'est moi qui vais retirer ma carte. C'est moi. Υπάρχει ένας παραπάνω από τους πρασίνους, αλλά θα βγάλω εγώ την κάρτα μου, εντάξει. Ωραία, είστε έτοιμοι. Πάμε. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 338. Α, όχι. Καταπίπτει. Συμβαστική 2β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. πολύ κοντά ήταν. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Συνεχίζουμε. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. καλησπέρα. Ε, ναι, είναι επειδή δεν σηκώνατε τα χέρια σας. Μην προσπαθείτε να το ρίξετε σε μένα. Πάμε κατευθείαν στην 446. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 4-2α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ποιος είπε ότι ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Δεν ήταν. «556. Υπέρ». Α, όχι, όχι, όχι, μάλλον. Ναι, μισό λεπτό. Ψηφίσαμε την 4-2α συμβαστική και είπαμε ότι απορρίπτεται. Ωραία. Επομένως, ναι, έχετε δίκιο. Παρακαλώ, το Λαϊκό Κόμμα. Ηρεμία. ψυχερεμία, όλα θα πάνε καλά. Απερίφθη λοιπόν η 4-2α. Γι' αυτό όντως θα ψηφίσουμε την 4-2 συμβιβαστική. Άρχεται η ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εντάξει. Τροπολογία 556. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική 4-3α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 4-3α. Non. Calmez-vous, ça va Ησυχία παρακαλώ, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 4-3α. Συμφωνεί. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην 558 σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα του 558. Πέρας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίζουμε από κοινού. Τις επόμενες τρεις ε, τροπολογίες. Υπέρ. Υπέρ. Κατά απορρίπτονται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 597. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το λογική σκέψη 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για την αιτολογική σκέψη 36. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 638. Α, όχι, καταπίπτει. 648 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 898 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει, άρχεται η ψηφοφορία για την 898. Πέρας. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 658 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 648. 88 συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 689. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Θέλετε να ελέγξουμε, εντάξει. Για την 689 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 518, τέταρτο εδάφιο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ας ψηφίσουμε. 518. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 518, πέμπτο εδάφιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 521. 721. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 721. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μικρή διαφορά. 744. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 518, 18 τρίτο εδάφιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9-2β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει, άρχεται. Η ψηφοφορία για την 9-2β. Πέρας. Ισοψηφία. Απορρίπτεται λοιπόν. Εννέα δύο αλφα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε χρονικά. Je ferme le vote. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οκτακόσια οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 794. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για τη συμβαστική 13. Υπέρ. Α, μισό λεπτό. Υπάρχουν ενστάσεις ως προς την προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε επί της ε, προφορικής τροπολογίας για το 13. Υπέρ. Κατά αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την προφορική τροπολογία για τη συμβαστική 13. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Et donc, L'amendement oral et le compromis 13 est adopté. Εγκρίνεται λοιπόν η προφορική τροπολογία και η συμβαστική 13. Πάμε στην 878. Υπέρ. 876, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, Αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 14. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση για αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Θα την ψηφίσουμε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ...923. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά εντάξει άρχεται πέρας απορρίπτεται Επιπρόσθετη ψηφοφορία για συμβαστική 14. Εδώ έχουμε μία σειρά τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Allez, je ferme Πέρας. Et c'est adopté. Εγκρίνεται. Καλά κάνατε και ζητήσατε επαλήθευση. 971. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 971. Άρχεται. Le vote est clos. Πέρας. Απορρίπτεται. 557 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15-2 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική 15.2 πέρας απορρίπτεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Να ψηφίσουμε τις πρόσθετες τροπολογίες. 989 και 990. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αυτές τις δύο τροπολογίες άρχεται. Je ferme le vote. Πέρας. Απορρίπτονται. 991. Ναι, προφορική τροπολογία, αν υπάρχει ένσταση, όχι. Ψηφίζουμε την τροπολογία σας, κύριε Μαρινέσκου, μην ανησυχείτε. Ελέγχω την κατάσταση. 991, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεν με εμπιστεύεστε κύριε Μαρινέσκου. Εντάξει, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Je Πέρας. Λυπάμαι κύριε Μαρινέσκου, αλλά απορρίπτεται. Allez, on va Πάμε τώρα στην προφορική τροπολογία για τη συμβαστική 17. Υπάρχουν ενστάσεις? Όχι. Ας ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα δώσω τη σκητάλη στον κύριο Μπούζεκ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Καριμά. Θαυμάσια τα πήγατε. Και τώρα προχωρώ στην συμβαστική 18. Υπέρ. 17 λέει η κυρία Αντελή. Πρώτα 17. Η κυρία Ντελή. Κυρίες και κύριοι, αν κοιτάξετε καλά την διαδικασία, θα δείτε ότι γράφει ότι προσθέτουμε προφορική τροπολογία στην συμβαστική 17. Επομένως, αν ψηφίσετε την προφορική, ψηφίζετε το συμβιβασμό που κρύβεται από πίσω. Άρα έχει εγκριθεί. Άρα προχωρούμε στην 18. Σας ξαναδίνω το λόγο, κύριε Μπούσεκ, για την προφορική τροπολογία 18. Δεν έχουμε και άλλη δυνατότητα παρά να ψηφίσουμε την συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «1002 υπέρ, συγγνώμη, 1012 κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά επαλήθευση επαλήθευση ε, κάποια ανάπαυλα χρειάζεται σας ευχαριστώ πέρα της ψήφου εγκρίνεται συμβαστική 27α υπέρ Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Πέρας. Απέριφθη. 22. Όχι, λέει κάποιος. Α, 22 λέει ο πρόεδρος ξεχωριστά. 22. Υπέρ, κατά, ας επαληθεύσουμε. Πέρας. Απερίφθη. 1074 υπέρ. Κατά. Νομίζω πρέπει να επαληθεύσουμε, δυστυχώς. 1074. Δύσκολο με δύο επιτροπές, λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Απερίφθη λοιπόν. Συμβιβαστική 28 με προφορική τροπολογία του Λαϊκού Κόμματος. Έχετε ενστάσεις πρώτα, πρώτα ενστάσεις. Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε ένσταση πρέπει να ηγερθείτε. Δεν χρειάζεται όμως. Ωραία. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78, 79, 80, 81. Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Όχι. Κάποιο λάθος. Περιμένω, περιμένω. Είστε έτοιμοι. Είστε όλοι έτοιμοι έτοιμες. 78 έως 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβαστική 3 3α υπέρ κατά ας ελέγξουμε επαληθεύουμε τη συμβαστική 3 εδάφιο 3α πέρας απορρίπτεται Συμβαστική 9, εδάφιο 4α. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε και εδώ. Συμβαστική 4α. Κλείνω την ε, ψήφο. Απεριφθεί. Συμβαστική 9, εδάφιο 4. Υπέρ, κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας επαληθεύσουμε. Πέρας. Εγκρίνεται βεβαίως. Συμβαστική 9, ε, 4α νέο, υπέρ, κατά Αποχές. Α, επαλήθευση. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3, 4β νέο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165. Υπέρ. Ας αρχίσουμε πάλι. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές, αλλά σε παληθεύσουμε, λέει ο πρόεδρος. Πέρας της ψήφου. εγκρίνεται. Ακολουθεί. 224. 224. Βρέστε το σας παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 233 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε 233 πέρα στη ψήφου εγκρίνεται 239 υπέρ κατά επαλήθευση 239 Πέρας. Απεριφθεί. 308. 308. Υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Πέρας. Απερίφθη. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε. Με ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται σαφέστατα. Συγχαρητήρια στους συγητές, όλους και όλες. Και ευχαριστώ πολύ την κυρία Πρόεδρο. Θαυμάσια συνεργασία μαζί σας κυρία Ντελή. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται για τον Δεκέμβριο του 2018. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Για τα μέλη της Ήτρε, σημαντικό. Έχουμε ακρόαση. Συνεχίζουμε τη συνάντησή μας στην αίθουσα 4Q2. Άρα όλοι και όλες μετακινούμεθα τώρα στην αίθουσα, αίθουσα 4Q2. Αρχίζει στις 10. Η Επιτροπή Μεταφορών παραμένει ωστόσο για να ψηφίσει εδώ, να συνεχίσει την ψηφοφορία εδώ, λέει η κυρία ε, Ντελή. Nous reprenons nos travaux. 10 και 30 επαναλαμβάνω τις εργασίες της Επιτροπής Μεταφορών στις 10 και 30 στην αίθουσα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Mes Κυρίες και κύριοι της Επιτροπής Μεταφορών, στην ημερήσια διάταξή σας λέει καθαρά ότι οι ψηφοφορίες προβλέπονται για τη ώρα 10 και 30. Κυρία Μέισνερ. Υπάρχουν και άλλοι τεχνικοί οι οποίοι φτάνουν στις 10 και 30. Το λέει στην ε, λίστα ψηφοφοριών, το λέει. Nous restons... Η Επιτροπή Μεταφορών παραμένει στην παρούσα αίθουσα. Αλλά επαναλαμβάνουμε τις εργασίες μας με ψηφοφορία στις 30. Το γράφει μέσα το έγγραφο που έχετε μπροστά σας.